Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Αν δεν καθίσατε ακόμα, παρακαλώ καθίστε. Καλώς ήρθατε στην έκδοση της εβδομάδας πόλεων και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετοί από εσάς ερχόσαστε από διάφορα μέρη. Θα υπάρξουν περίπου 7.000 άνθρωποι εδώ, στις Βρυξέλλες, για να παρασταθούν σε αυτή την εκδήλωση αυτή την εβδομάδα. Θα είναι πολύ άσχολη η ατζέντα, πολύ άσχολο το πρόγραμμα και γι' αυτό δεν θέλουμε να χρονοτριβούμε και ξεκινάμε αμέσω. Πριν μπούμε στην καρδιά του θέματος και πριν συζητήσουμε το πώς οι πόλεις και οι περιφέρειες αποτελούν τους πυλώνες του μέλλοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να αναφερθώ σε κάποια διαδικαστικά Καταρχάς παρακαλώ ε, να βουβάνετε τα τηλέφωνά σας και μην τα σβήσετε γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα τηλέφωνά σας σε λίγο. Απλώς χωρίς ήχο να τα έχετε. Θα κάνουμε κάποιες ε, βολιδοσκοπήσεις ε, σε αυτή τη συνεδρίασή μας και θα θέλαμε να μπορείτε να συμμετάσχετε με τα τηλέφωνά σας. Παρακαλούμε επίσης και να βάλετε μηνύματα στο Twitter. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, σε όλη αυτή την εβδομάδα, θα ενδιαφερθούν. Και αν δεν καταφέρουμε αυτή η εκδήλωση να γίνει ε, δημοφιλής εκδήλωση, δεν θα κάνουμε πολύ καλά. Λοιπόν, έχετε, θα έρθει και το hashtag, θα το δείτε, ε, ανεβάστε μηνύματα στο Twitter, EU Regions Week. Έχουμε διαρμηνία σε 24 γλώσσες. Διαλέξτε το κανάλι σας, δεν θα σας ε, παριθμίσω όλα τα κανάλια. Διαλέξτε το κανάλι της επιλογής σας για να μπορέσετε να ακούσετε τη διερμηνία στη γλώσσα σας. Επίσης είμαστε στο διαδίκτυο μέσω web streaming. Χαιρετίζουμε λοιπόν όλους που μας παρακολουθούν από διάφορα μέρη, από τα σπίτια τους, από τα γραφεία τους, τους τοπικούς, πολιτικούς, περιφερειάρχες κλπ. που δεν μπορεί να είναι εδώ. Ελπίζουμε να απολαμβάνετε αυτή την εκπομπή και καλείστε να θα κληθείτε στο slider να συμμετάσχετε στις διάφορες βολιδοσκοπήσεις που θα κάνουμε. Όπως ξέρετε, θα είναι δύσκολη εβδομάδα και συνεδρίαση δύσκολη. Θα, θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Θέλουμε να είμαστε πολύ διαδραστικοί. Αλλά με 900 άτομα στην αίθουσα θα είναι δύσκολα. Θα κάνουμε όμως ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τηρήσουμε το πρόγραμμα. Είναι και δύσκολε οι πολιτικέ εποχέ που περνάμε. Έχουμε ένα νέο Ευρωκοινοβούλιο, όπω ξέρετε. Σύντομα θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε νέα Προέδρο, υπερχόμενη Προέδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και έχουμε ένα νέο πολιτικό πρόγραμμα για όλους μας και για σας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτή την εβδομάδα Πρέπει να δούμε πώς μπορείτε εσείς να συμβάλλετε, να παίξετε το ρόλο σας, να ενισχύσετε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πώς αυτές υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Πώς μπορείτε κι εσείς να προωθήσετε το ευρωπαϊκό ιδεώδες στο δικό σας επίπεδο. Θα εξασφαλίσουμε το ότι αυτή η εβδομάδα είναι δική σας Κυρίω στην υλοποίηση του προγράμματο και στην οργάνωση του προγράμματος αυτό φροντίσαμε. Ελπίζω να το απολαύσετε το πρόγραμμα και να χρησιμοποιήσετε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει. Για να το κάνουμε αυτό θέλουμε σήμερα να επικεντρωθούμε επί τριών βασικών θεμάτων. Αυτά καθ' αυτά τα θέματα καλύπτουν και άλλα θέματα προ συζήτηση που θα συζητηθούν αυτή την εβδομάδα. Τα βασικά θέματα για σήμερα είναι η αλληλεγγύη πώς μπορούμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτει περισσότερους ανθρώπους, πιο συμπεριληπτική, βιωσιμότητα, αλλαγή του κλίματος. Κάνουμε αρκετά, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Τι κάνουμε ακριβώς και τι αντίκτυπο έχουν αυτά που κάνουμε. Και τέλος, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πλησιάσει τους πολίτες της. Αυτό το βλέπουμε συχνά μπροστά μας στα θέμα, πολλοί από εμά το εξετάζαμε, προβληματιζόμαστε, το επεξεργαζόμαστε επί σειρά ετών. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω προσωπικά ότι ένα κομμάτι της απαντήσεως είναι στα χέρια σας, παιδιά, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για να το καταφέρουμε αυτό, έχουμε εντυπωσιακό κατάλογο μιλητών. Πρώτα απ' όλα, την κυρία Κλάρα Ντόμπρεφ, που μας φιλοξενεί, που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Παϊκού Κοινοβουλίου που είναι υπεύθυνη για τη σχέση με την Επιτροπή των Περιφερειών μεταξύ άλλων. Η κυρία Ντόμπρεφ παρακαλώ να έρθει. Κύριος Καλ Χάινς Λαμπέρτ, Πρόεδρος Επιτροπής των Περιφερειών, παρακαλούμε να έρθει εδώ. Η κυρία Σμπιέτα Μπιενκόφσκα, Ευρωπαία Επίτροπος που είναι υπεύθυνη για την ενία αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. και για να του κρατήσει παρέα να τους κρατήσουν παρέα έχουμε πέντε εκλεγμένα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης Λάρας Παραβινιέρα Δημοτική Σύμβουλος στο, στη Φλωρεντία, στην Ιταλία Βερσόν Σοβέ Δήμαρχος της Οτάν στη Γαλλία Μία Εσκελίνεν Φιγκερός, δημοτική σύμβουλος από το Κουόπιο, από τη Φιλανδία. Η κυρία Κέρστιν Κάρι, σύμβουλος στο Συμβούλιο του Highlands στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και τέλο Ράτος Φαλσφόλ, δημοτικός σύμβουλος στο Μιέλετς στην Πολωνία. Καλώς ήρθατε όλοι. Είπα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να είμαστε διαδραστικοί. Λοιπόν, βγάλτε τα τηλέφωνά σας. Θα έχουμε μια ερώτηση για το Slido. Συνδέστε με το slido.com Slido Do, ότι είναι πιο εύκολο για εσάς να συνδεθείτε. Βάλτε το hashtag EU Regions Week. Να σας δώσω ένα λεπτάκι να συνδεθείτε. Εσείς που μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο, παρακαλώ κάντε το ίδιο. Μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συνεδρίαση. Παρακαλώ να ψηφίσετε. Εντάξει. Slido.com μπήκατε. EU Regions Week. Μάλιστα. Και η ερώτηση θα εμφανιστεί. Δύσκολο να διαβάσετε μεγάλη οθόνη, αλλά υπάρχει λόγος. Γιατί θέλουμε να κοιτάξετε τις οθόνες από τα τηλέφωνά σας για να ψηφίζετε. Η ερώτηση αφορά τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Το Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal, μια οικονομία που είναι για τον κόσμο, ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο, μια Ευρώπη που μπορεί να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή ή να αφορά την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής η Ευρώπη. Να σας δώσουμε ένα λεπτάκι και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ψηφίσατε όλα ξεκάθαρα. Η τάση φαίνεται να σταθεροποιείται. Λοιπόν, πού καταλήγουμε, το ευρωπαϊκό Green Deal κερδίζει τις περισσότερες ψήφους. Και μετά ακολουθεί με μικρή διαφορά μια οικονομία που τελικά έχει αποτελέσματα για τον κόσμο και αυτές οι δύο τάσεις προηγούνται των άλλων. Νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει ένα από τα θέματα των συζητήσεών μας σήμερα το απόγευμα. Αναφέρθηκα στη βιωσιμότητα και ότι θα συζητήσουμε και την αλλαγή του κλίματος όπως σας είπα. Το πρώτο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε που σχετίζεται με το πώς η οικονομία μπορεί να δώσει αποτελέσματα στον κόσμο είναι η αλληλεγγύη. Και γι' αυτό θα ήθελα να στραφώ προς τον πρώτο, στην πρώτη ομιλήτριά μας, τη Λάουρα Σπαραβίνια. Λάουρα, είσαι δημοτική σύμβουλος στη Φλωρεντία, αλλά ασχολείσαι και με κοινωνικά θέματα, είσαι κοινωνική λειτουργός. Πόσο νομίζει ότι η πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τη διαφορά, Πόση διαφορά νομίζει ότι έχει κάνει όσον αφορά την πόλη σου Ποια πρέπει να είναι η προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, σοφά τη συνοχή, κατά την άποψή σου. Καταρχά, να ευχαριστήσω όλου σα που μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι εδώ. Λοιπόν, έχουμε με κήπο, το Τζαντίνο Δεκαζόμετρο. Εκεί υπάρχουν διάφορε υπηρεσίε όπω είναι πιαγωγείο, διάφορα κέντρα με ανθρώπους που έχουν ψυχικά προβλήματα για θέματα υγείας. Λοιπόν, στη Φλωρεντία λοιπόν αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των προβλημάτων ανοίγοντας αυτό το κέντρο που ήταν δημοφιλές. Ένα, μια ταβένα, ένα, ε, ένα εστιατόριο. θα πρέπει να έγινε μια προσέγγιση που καλεί τους πάντες. Ε, πρόνοια που φέρνει τους ανθρώπους κοντά μας σε επαφή με άλλους μέσω της συνύπαρξης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον και να δούμε ποια είναι δύναμη του ανθρώπου. Την δύναμη που έχει η διάδραση μεταξύ των ανθρώπων που επιτρέπει στον άλλον να μην αισθάνεται ότι είναι ξένος εχθρός αλλά ο άλλος είναι κάποιος που μπορεί να μας βοηθήσει, που μας ενισχύει αν μπορούμε να ε, έχουμε μια ενσυναίσθηση απέναντί του. Άλλο ένα παράδειγμα. Ένας, ένας γέρος που διαβάζει στα παιδιά των μεταναστών παραμύθια. Αυτό βλέπουμε το παιδί ότι είναι ένα παιδί, δεν είναι κάποιος που πρέπει να τον αποφύγουμε. Ένταξη είναι το μυστικό. Είναι η βάση της συνεργασίας η ένταξη. Έτσι, οι κοινωνικές πολιτικές λειτουργούν σαν το ράφτη που σειράπτει τα κομμάτια της κοινωνίας και δημιουργεί μια κοινή πρόνοια ε, όπου όλα λειτουργούν. Και αυτό ήθελα να σα πω, αυτό το μοντέλο να παρουσιάσω. Δηλαδή κινητήρια δύναμη για την ευημερία, την πρόνοια. Όλοι συνεργάζονται και εμπνέονται από την ευημερία τη κοινωνία. Και ο καθένα εμπνέεται από τι δυνατότητε που έχει, τι μπορεί να προσφέρει. Και ανάλογα με την ηλικία του προσφέρει. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εδώ βρισκόμαστε και θέλω να, με, διαβιβάσω τι κάνουμε στη χώρα μου. Αλλά θέλω να έχουμε και κοινό τόπο συζητήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα, όπως ε, συγγνώμη, είμαι λίγο ταραγμένη. Το θέμα της ε, αλλαγής του κλίματος, Φερρυπίν. Ε, το δημογραφικό πρόβλημα, ψηφιακή επανάσταση που αλλάζει την αγορά εργασίας. Έχουμε προβλήματα και έχω μία ερώτηση για όλους μας εδώ που θα συζητήσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σταθούμε στα πόδια μας, να αντιμετωπίσουμε αυτά. Διότι αυτό είναι το θέμα για το μέλλον. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα ετοιμάσουμε ένα έγγραφο πολύ ενδιαφέρον που δεν θα έχει νόημα. Θα επιστρέψω κι εγώ στη χώρα μου διαφορετικά, θα αντιμετωπίσω του πολίτε μου και δεν θα έχω απάντηση για αυτούς και θέλω να έχω απάντηση για τους συμπολίτε μου. Λοιπόν, επειδή ε, είμαι δημοτική σύμβουλος και κοινωνική λειτουργός, θέλω να βρίσκω συγκεκριμένε απαντήσεις και έχω κάτι που θα συζητήσω μαζί σας. Θα μπορούσαμε, ίσως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκό σύστημα πρόνοιας. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πρόνοιας θα ήταν η μόνη στρατηγική για να φροντίσουμε κάθε πολίτη σε όλη την ένωσή μα, χωρίς να υπάρχει διαφορά, χωρίς να έχει, υπάρχει ασημετρία επαγγελματική ή μισθολογική. Λοιπόν, βλέπετε, είμαι, ε, πάντα μελετούσε αυτό το θέμα και ε, επειδή τα αισθάνομαι αυτά τα θέματα στην καρδιά μου, γι' αυτό μπερδεύομαι και μεταραγμένη. Ξέρω ότι έχουμε την απάντηση για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε η δύναμή τους. Μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουν συνεργαζόμενοι. Βασικός στόχος της ευρωπαϊκής πρόνοιας θα ήταν όλοι μαζί να βρούμε κοινά πρότυπα κάθε ένας τοπικός πολιτικός θα μπορέσει να υλοποιήσει την πολιτική. Πώς, χάρη σε τι, χάρη σε εμάς, χάρη στην πολιτική συνοχής, στις πολιτικές συνοχής, χάρη στη σωστή διακυβέρνηση, χάρη στην επικουρικότητα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα της ευρωπαϊκής πρόνοιας, να διαμορφώσουμε την αγορά εργασία, ώστε να μπορούμε να συγκεράσουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ας ξεκινήσουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος προνοίας, να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα κοινωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα σύστημα οικονομικό και σύστημα απασχόλησης. Οι κοινωνικές πολιτικές είναι η μόνη δύναμη και το μόνο πράγμα το οποίο εμείς σαν πολιτικοί μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να πετύχει την κοινωνική δικαιοσύνη, ο κόσμος να μπορεί να πετύχει ισότητα. Ε, ε, πρόνοια δεν είναι απλώς ένα στοιχείο του προπολογισμού, αφορά τις επενδύσεις, αφορά το να λάβουμε υπόψη ότι ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Λάουρα. Πολύ παθιασμένη ομιλία και πολύ ωραίος τρόπος να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Τώρα να στραφώ στο δεύτερο συμμετέχοντα στο πάνελ, στον ε, Μύροσλαβ. Μύροσλαβ, ποια ήταν μεγαλή, ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της, του Δήμου σας. Ποια ήταν η νούμερο ένα προτεραιότητα για σας. Ακούσαμε τη Λάουρα. Εσείς τι θα είχατε να μας πείτε. Ευχαριστώ. Αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα, παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας, Νομίζω πρέπει να με ακούτε από το κανάλι 18. Αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα και είναι αντιληπτό σε όλους είναι οι υποδομές σε οδικά δίκτυα, σιδηροδρόμους, ε, τις υποδομές των μεταφορών καθώς και τις σωστές διασυνδέσεις. Εγώ ζω στα νοτιοανατολικά της Πολωνίας και είμαστε πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο Α4 που συνδέει την ανατολική πλευρά της χώρας με τη δυτική προς τα δυτικά σύνορα. Τα ανατολικά μας σύνορα είναι και ανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ λοιπόν ήρθα στις Βρυξέλλες ξεκινώντας από ένα τοπικό αεροδρόμιο στην πόλη της Γιασόνκα, στην δική μου την περιφέρεια. Το αεροδρόμιο αυτό περνάει μια φάση εξυγχρονισμού τώρα με ευρωπαϊκά κονδύλια και ένα άλλο σημαντικό έργο υποδομής είναι ένας άλλος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει τις χώρες της Βαλτικής μέσω της Πολωνίας με τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και θα φτάνει και ως την Ελλάδα. Είναι η λεγόμενη Καρπαθία Οδός. Εάν σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όντως να εξαλείψει τα σύνορα στην Ευρώπη, ε, αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με γραφειοκρατικό τρόπο. Πρέπει να υπάρξουν και διασυνδέσεις υλικές, απτές, χειροπιαστές. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, συνοχή. Η συνοχή και εδώ είναι πολύ σημαντική, αλλά και τα κονδύλια συνοχή είναι σημαντικά για τη χώρα μου, όπω τα γνωρίζετε. Ε, κάτι που πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να δώσουμε μια νέα όθηση στην έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία και να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση, ιδίω στου τομεί που θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε νέα προστιθεμένη αξία, νέες λύσεις για το περιβάλλον, για την προστασία του περιβάλλοντος. Πολλά κράτη-μέλη έχουν διαφορετικό, δυναμικό και πολλές φορές και ανεκμετάλλευτο. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε και στους νέους μια ευκαιρία να δείξουν ε, τις δυνατότητές τους σε όλο τους το μεγαλείο. Στις χώρες τους ε, και ιδίως στις χώρες προέλευσής τους, χωρίς να χρειάζεται να μεταναστεύσουν να μετακινηθούν. Ε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε περιοχές του κόσμου όπως η Κίνα ή οι Ηνωμένε Πολιτείε στο μέλλον. Διότι πίσω από κάθε εφεύρεση, πίσω από κάθε καινοτόμο λύση βρίσκεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο. Ε, αυτοί οι άνθρωποι ε, σήμερα δεν μπορούν να πετύχουν κάτι ιδιαίτερο χωρίς θεσμική στήριξη. Αυτή την κατεύθυνση πιστεύω πρέπει να ακολουθήσουμε νέες ιατρικές λύσεις, νέε τεχνολογικές λύσεις, προστασία του κλίματος. Αυτές είναι οι προκλήσεις που χρειαζόμαστε ε, να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Εάν διοχετεύσουμε την ενέργειά μας στις σωστές κατευθύνσεις μπορούμε να ζήσουμε και περισσότερο και να ε, δωρήσουμε έναν υγιή πλανήτη στις επόμενες γενιές. Σε ευχαριστούμε πολύ Ράντοσλαβ. Πριν δώσω το λόγο στους τρεις θεσμικούς μας ομιλητές για να απαντήσουν στις εκκλήσεις και τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Ήθελα να καλέσω ένα από τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών να ε, μας εκφράσει και εκείνη την έκκλησή της. Κυρία Ζαμπέλ Μπουντινό, παρακαλώ, μπορείτε να απευθυνθείτε στους συμμετέχοντες του πάνελ. Κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο αυτό πάνελ αφιερώθηκε στο θέμα της αλληλεγγύης, ενώ το δεύτερο αφορά την βιώσιμη Ευρώπη. Βλέπουμε ότι τα περιβαλλοντικά θέματα ε, είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους εδώ. Ήθελα να πω ότι μετά την μελέτη για την ε, ανισότητα ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον, οργανισμό, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος έχουμε πλέον και στατιστικά δεδομένα για να δούμε ότι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες κοινωνικές δυσκολίες και τις μεγαλύτερες ανισότητες είναι αυτές που είναι και περισσότερο εκτεθειμένες στις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζητούμε από τους πολίτες και τις διάφορες περιφέρειες ιδιαίτερες προσπάθειες όταν είναι αυτοί που περισσότερο και σε σύγκριση με τις πλουσιότερες περιοχές. Γι' αυτό αυτό χαίρομαι για την πρόταση της κυρίας Φοντερ Λάιεν για μια νέα πράσινη λύση για την Ευρώπη, αλλά δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί. Θα πρέπει να μην πληγεί η πολιτική της συνοχής. Θα πρέπει να γίνουν και κρατικές επενδύσεις στις περιφέρειες που έχουν δυσκολίες και βρίσκονται σε υποβάθμιση. Καταπολεμώντας κοινωνικές υπερβολοντικές δυσκολίες και ταυτόχρονα προστατεύοντας το περιβάλλον. Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι η τοπική, αυτή που λαμβάνει υπόψη τι τοπικέ ιδιαιτερότητε. Και έτσι προκύπτει ένα διπλό ερώτημα. Πώ μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι τα χίλια δι ευρώ για την οικολογική μετάβαση που προβλέπονται ω επένδυση μπορούν να επενδυθούν με τοπικό χαρακτήρα, με τοπικά κριτήρια. Και πώ μπορούμε να διακρίνουμε τι περιβαλλοντικέ πολιτικέ από το πρόγραμμα Juncker και το InvestEU, που πιο πολύ σκοπό έχουν να παράγουν προγράμματα για ιδιαίτερα ανταγωνιστικέ περιοχέ ε, κυρίως και πρωτεύουσες Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω έχουμε πολλά που μπορούν να μας απασχολήσουν και γι' αυτό θα ήθελα να στραφώ στην κυρία Ντόμπρεφ για να δώσει πρώτη κάποιες απαντήσεις. Η κυρία Ποντινό ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο και για το δεύτερο θέμα, το δεύτερο πάνελ που θα μας απασχολήσει σήμερα αν θέλετε όμω να απαντήσετε και στου δύο πρώτου ομιλητέ και εν μέρη και στο σχόλιο τη κυρία Μπουντινό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που είστε εδώ και που με καλέσατε κιόλα. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα. Η πολιτική συνοχή είναι μια μοναδική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αποδείξει τα αποτελέσματά τη τι περασμένε δεκαετίε. Δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται αλλαγέ, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται βελτιώσει, αλλά το σημαντικό είναι να τη διατηρήσουμε και να αγωνιστούμε ώστε η χρηματοδότηση να μην μειωθεί το ερχόμενο διάστημα προγραμματισμού, δημοσιονομικού προγραμματισμού. Η πολιτική συνοχή είναι αλληλεγγύη. Σημαίνει αλληλεγγύη μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών, ευρωπαϊκών περιφερειών και περιοχών. Αυτό είπε ο Ράντοσλαβ στην ουσία. Ε, τι είδου επενδύσει στι υποδομέ χρειαζόμαστε για να αναβαθμίσουμε τι περιοχέ που να μην, μπορεί να μην έχουν τόσου πόρου όσο οι άλλε. Ε, και η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και των περιφερειών ήταν η κατευθυντήρια γραμμή, ήταν η πηξίδα και ο, ο στόχο προ τον οποίο όδευε η πολιτική συνοχή τα τελευταία χρόνια. Πρέπει λοιπόν να φουγκραστούμε και τι δικέ σα απόψει. Γι' αυτό παροτρύνω ε, όλου και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι η μελλοντική περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού και από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι με 500 ε, εκατομμύρια πολίτε μια έκφραση αλληλεγγύη. Πρέπει να πάμε πιο μακριά. Πρέπει να πάμε ε, παραπέρα. Ε, αλληλεγγύη με του καθημερινού πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να δούμε. Αλληλεγγύη σημαίνει να αντιμετωπίσουμε τα δικά του, δικά της ε, ή τα δικά του προβλήματα ε, ως προς την κοινωνική κάλυψη, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση μην έρχεστε να δημιουργήσετε ένα ψευδό δίλημα ότι το πρόβλημα είναι ο ανταγωνισμός σε αντιδιαστολή με την με την εκπαίδευση. Έχουμε κόσμο ο οποίος είναι μορφωμένος και ζει σε ανασφάλεια. Οι χώρε όμω είναι πλέον ανταγωνιστικέ, είναι αυτέ που έχουν υψηλή εκπαιδευτικό επίπεδο και στέγαση για του πολίτε του. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν πού ε, υπάρχουν διαφορέ και πώ θα προωθήσουμε το δεύτερο πυλώνα τη αλληλεγγύη, ε, δηλαδή την κοινωνική Ευρώπη. Αυτό θα πει για μένα ο δεύτερο πυλώνα. Εν μέρει έχουμε κάποια εργαλεία και εντό τη πολιτική συνοχή. Την εγγύηση για τα παιδιά, για την οποία έχουμε πιέσει πολύ, α πούμε. Ή το πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων. Αλλά πρέπει να αναπτύξουμε πολύ περισσότερο την πολιτική αυτή. Και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε στην πολιτική συνοχή, ιδίω για κοινωνικά ζητήματα, πρέπει να αποφασίζονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον κόσμο, στους ανθρώπους. Τα κονδύλια και οι πόροι να πάνε κοντά στους πολίτες. Διότι κανείς άλλος δεν ξέρει τόσο καλά τι χρειάζονται εδώ στις Βρυξέλλες ε, οπουδήποτε για το τι χρειάζονται καθημερινοί αυτοί άνθρωποι. Ε, η Λάουρα και εγώ τα ξέρουμε καλά. Ε, και ναι, χρειάζονται νέε δεξιότητε, νέε διαδικασίε. Ευχαρίστω να μα απασχολήσει ω θέμα το, ε, τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, τα ελάχιστα υγειονομικά πρότυπα, τα ελάχιστα εκπαιδευτικά πρότυπα και ο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα ζητήματα που μα χρειάζονται. Διότι κοιτάξτε μα λιγάκι, καθόμαστε εδώ σε μια από γοργότερα αναπτυσσόμενε οικονομίε στον κόσμο. Καθόμαστε σε μια από τι ε, ευπορότερε κοινωνίε του κόσμου. Είμαστε στον 21ο αιώνα και μιλάμε για παιδική φτώχεια. Μιλάμε για κόσμο που δεν έχει κανονικό κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Πραγματικά δηλαδή, τι κάνουμε. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό, θα έρθουν άλλα προβλήματα. Λαϊκισμοί, εξτρεμισμοί, και θα δούμε τι θα ακολουθήσει και το Brexit. Δεν θέλω καν να το φαντάζομαι. Η αλληλεγγύη λοιπόν αυτό είναι για μένα και είναι η στόχη για το μέλλον. Ευχαριστούμε κυρία Ντόμπρεφ. Επίτροπε Μπιενκόφσκα. Θέλετε να μας πείτε και εσείς τις απόψεις σας. That's okay. Works as well. Okay. <laughs> Uh, so... Μπορείτε και έτσι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τις ευχαριστήσεις, που θέλω να στείλω στην Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο και να σας πω πως είμαι υπεύθυνη για την ενιαία αγορά τώρα και για τα τελευταία 20 χρόνια της ε, ε, ζωής μου ήμουνα και εγώ στην ε, διεύθυνση για την περιφερειακή πολιτική και βλέπω πολλούς φίλους εδώ στην αίθουσα και είναι πραγματικά εντυπωσιακή αυτή η εκδήλωση που μας επιτρέπει να συζητήσουμε τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με τον διάλογο, τις κοινέ λύσεις, τους κοινού τόπους. Πολλά έχουν υποθεί ήδη Και επειδή τα τελευταία πέντε χρόνια ασχολούμαι με την ενιαία αγορά, να σας πω πως δεν είναι τυχαίο πως η συνθήκη της Ρώμης έστησε την ενιαία αγορά και μετά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Γιατί αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής είναι πολιτική αλληλεγγύης και δι εσείς που είστε σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, εφαρμόζετε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές επιτόπου και οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ή εθνική πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες και η πολιτική συνοχής είναι πραγματικά μία μοναδική πολιτική όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίω. παρόλο που και σε άλλα σημεία της οικουμένης είδα να υπάρχουν τέτοιου είδους προσπάθειες δηλαδή δημιουργία κάτι παρόμοιο με την πολιτική συνοχής. Εγώ ερωτεύτηκα την πολιτική αυτή πολλά χρόνια πριν είναι κάτι το πολύ δημοφιλές σήμερα είναι μια ολιστική, για να την πω έτσι, πολιτική με οριζόντιες λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και πολλές τοπικές κυβερνήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μεγάλες υποδομές, με τις επενδύσει. Μας μιλήσατε για τον αυτοκινητόδρομο Α4 στην Πολωνία και άλλοι αυτοκινητόδρομοι και οδικοί άξονε, που ήταν δικό μου σχέδιο τότε γιατί ήμουνα υπουργό ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης και μετά περνάμε σε στόχους παιδείας, εκπαίδευσης και φτάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο που συμπληρώνει τα υπόλοιπα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, όσο γίνεται. Επειδή είμαι επίτροπο τη ενιαία αγορά, να σας πω πω βεβαίω και δεν χρησιμοποιούμε το πλήρε δυναμικό τη ενιαία αγορά. Η πολιτική συνοχή και η απόλυτα πλήρης ενιαία αγορά θα μπορούσαν να μας μετατρέψουν στον πιο σκληρό ανταγωνιστή των φίλων μας σε άλλες αγορές όπως η Κίνα, η ΕΠΑ και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά λοιπόν τα δύο εργαλεία θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και ακολουθώντας τις πολιτικές μας γιατί η πολιτική συνοχής κάποιος το είπε είναι μια πολιτική που μεταλλάσσεται με το χρόνο Είδαμε το Green Deal και είδαμε και την πρωτοβουλία πολίτες, Ευρώπη για τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα εργαλεία να τα χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο και αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές. Σας παρακαλώ λοιπόν, χρησιμοποιήστε αυτές τις λίγες μέρες που έχετε στη διάθεσή σας. Και μην μιλάτε μόνο για τις καλύτερες πρακτικές αλλά και για τις χειρότερες. Συζητήστε με τους φίλους σας που κάνατε λάθος, που αποτύχατε γιατί αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει αυτά τα δύσκολα ζητήματα να τα αντιμετωπίσουμε και έχουμε να απαντήσουμε και πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Προτεραιότητες, το Green Deal, πώς θα είναι. Επίσης, και νομίζω ότι αυτό θα δώσει μια μετάβαση στην επόμενη συζήτηση που είναι αυτή της βιωσιμότητας, αλλά θα πρέπει να προσφέρουμε στους πολίτες μας αυτό που μας ζητούν και αυτό δεν συνέβαινε πριν από 5 και 10 χρόνια το βλέπουμε όμως και από το τι ψηφίζουν αυτό θέλουν οι Ευρωπαίοι αυτό ζητάνε Γι' αυτό κατεβαίνουν στον δρόμο. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και τα στόματά μας και να πούμε όχι δεν υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν και είναι κορυφαίες προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους πολίτες και θα τα καταφέρουμε. Και ίσως αργότερα να ξαναπάρω το λόγο για να πω δύο λόγια, αλλά η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική την οποία θα πρέπει να φροντίσουμε, να τη συζητήσουμε, να την αλλάξουμε, αλλά είναι μια μοναδική πολιτική και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, στο έπακρο. President ο πρόεδρος Λάμπερτ, τι έχετε να πείτε εσείς για να βελτιώσουμε ή για να διαδώσουμε πιο πολύ την πολιτική συνοχή. Είναι η 17η φορά που εορτάζουμε αυτή την εκδήλωση και έρχεται σε μια στρατηγική στιγμή. Έχουμε νέα θητεία στο Κοινοβούλιο, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πολλές προκλήσεις. Τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα, θα τα αλλάξουμε όλα? Πολλά, ναι, θα πρέπει να αλλάξουμε. Αλλά θα πρέπει επίσης να έχουμε συγκεκριμένους στόχους και να γνωρίζουμε πώς θα τους πετύχουμε. Πιστεύω πως ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών και το να τοποθετήσουμε σωστά την Ευρώπη μέσα σε ένα κόσμο που συνέχεια αλλάζει. Πρέπει να έχουμε ισχυρά θεμέλια οικονομικά, πολλά έχουμε κάνει, αλλά κανείς δεν έχει κατακτήσει το τέλειο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε εξίσου στέρεα θεμέλια οι πυλώνες στο κοινωνικό κομμάτι. Γιατί είμαστε μία ήπειρος πολύ πλούσια είναι απαράδεκτο λοιπόν ένα τέταρτο του πληθυσμού να διαβιώνει πολύ κοντά στο κατόφλι της φτώχειας. Πάρα πολλά μένουν να γίνουν και αναφερθήκατε και στις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει από την Ιταλία. Τι είναι όμως το πιο σημαντικό. Είναι η μέθοδος που θα ακολουθήσουμε. Η πολιτική συνοχής, την οποία κάποιοι χαρακτηρίζουν ως απαρχαιωμένη πολιτική, είναι το εργαλείο του μέλλοντος. Και τούτη τη βδομάδα εμείς αποδεικνύουμε πως αυτό ισχύει. Η πολιτική συνοχής είναι αυτή όπου το τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να συνεργαστούν έτσι ώστε να πετύχουν στόχους που έχουν θέσει. Είναι η μόνη πολιτική που υπάρχει αυτή η τέλεια ισορροπία και γι' αυτό θα πρέπει να την στηρίξουμε, να την αξιολογήσουμε, να την αναμορφώσουμε αλλά κυρίως να την αγκιστρώσουμε στους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Χρειάζεται λοιπόν να κινητοποιηθούμε. Χρειάζεται όλοι σε τοπικό επίπεδο να συνεργαστούν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβολίου, ο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 761 βουλευτές, οι 10.000 εθνικοί βουλευτές στα κράτη-μέλη και το 1 εκατομμύριο ερετών στην τοπική αυτοδιοίκηση, για να σας εξηγήσω τα νούμερα όλοι αυτοί πρέπει να κινητοποιηθούν υπέρ των στόχων στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται για το μέλλον της Ευρώπης. Και όσοι θέλουν να κινδυνεύσει η Ευρώπη να μην καταφέρουν τίποτα. Είναι λοιπόν η εβδομάδα αυτή των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων μια τεράστια ευκαιρία για να συνεργαστούμε και να τα πάμε καλύτερα στο μέλλον. Νομίζω ότι καλά ξεκινήσαμε. Πολύ συγκινητικές εκκλήσεις για βελτίωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Και αν απολαύσατε αυτή τη συζήτηση και ο πρόεδρος Λάμπερτς απέθυνε έκκληση σε όλους σας σε όλους τους ντόπιου πολιτικούς να δραστηριοποιηθούν. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω συμμετοχής στην συμμαχία μας της συνοχής Είδα κάποια δημοσιεύματα, έξω, κάποια έντυπα που περιγράφουν αυτή τη συμμαχία. Αν δεν ρίξατε μια ματιά, κάντε το. Δείτε τα διάφορα έντυπα και στο hashtag Cohesion Alliance παρακολουθήστε το ιστορικό και γίνετε μέλη της, της συμμαχίας για τη συνοχή. Μιλήσαμε για κοινωνική συνοχή. Εκεί τίθε το θέμα της βιωσιμότητας και της αλλαγής του κλίματος. Είναι κεντρικό θέμα δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς, αλλά όπως είπε και την πρόεδρος Ντόμπρεφ, είναι κάτι που αφορά όλους τους πολίτες μας. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να σκεφτούμε τη διάσταση της βιωσιμότητας όταν μιλάμε για αλληλεγγύη. Το ανέφερε η κυρία Μπουντινός. Στρέφουμε τώρα προς το επόμενο, στο Βινσάν Σοβίτ, το επόμενο μέλος του πάνελ που είναι ο δήμαρχος τότε στη Γαλλία, Βανσάν. Ξέρουμε, αντιμετωπίζουμε κάτι που δεν είναι καν κρίση, είναι κατεπίγουσα ανάγκη και είναι πρόβλημα, είναι πρόκληση. Πρέπει να μειώσουμε τι συνέπειε της αλλαγή του κλίματος και μετά να προθίσουμε τη συνοχή και την αλληλεγγύη. Η κυρία Ντόμπρεφ είπε ότι ίσως δεν είναι συζήτηση. Δεν θέτουμε το ένα θέμα εναντίον του άλλου. Κατά την άποψή σα όμω, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πρέπει να κάνει για να βοηθήσει τις πόλεις και τις περιφέρειες να μειώσουν τις συνέπειες αυτών των φαινομένων και να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος, από τη δική σας εμπειρία. Κάνουμε αρκετά. Ευχαριστώ Φλωρόνς για την ερώτησή σου πολύ ευρεία. Σε ένα τρίλεπτο θα προσπαθώ να δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα βασιζόμενο σε αυτά που είπε πρόεδρος, ο πρόεδρο τη Επιτροπή των Περιφερειών. Πώ μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με την τοπική αυτοδιοίκηση για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματο και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαι δήμαρχο μια πόλη που έχει 14.000 κατοίκου κοντά στο Μορβά, στην περιοχή του Μορβά και έχουμε δάση, 40% της, του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ενώσης καλύπτει από δάση. Και όμως τα δάση δεν αναφέρονται εντός των συνθήκων και η δασική πολιτική είναι σε, ε, ακόμα σε αρχικό στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει σημαντική δουλειά. Κάθε φορά αναλύεται και αναθεωρείται αυτή η στρατηγική και υπενθυμίζεται η σημασία που έχουν τα δάση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά πώς μπορούμε να μειώσουμε τα αποτέλεσματα της αλλαγής του κλίματος, να καταπολεμήσουμε ε, την άνοδο της θερμοκρασίας και τις αρνητικές συνέπειες της απώλειας της βιοπικιλότητας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την πολιτική των δασών. Σήμερα αυτός ο τομέας είναι κάπως εγκαταλελειμμένος, είναι στα χέρια των κρατών μελών και πολλά κράτη-μέλη δεν διαχειρίζονται με βιώσιμο τρόπο τα δάση. Πώς μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε πιο μακριά και είναι θέμα και κοινωνικό αυτό, διότι στη δασική εκμετάλλευση πολύ συχνά έχουμε και εκμετάλλευση των εργαζόμενων στη δασοκομεία που ε, είναι ε, εργαζόμενοι που είναι αποσπασμένοι, είναι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζονται σε τραγικές συνθήκες. Εργάζονται εκεί που δεν θέλουν πλέον οι, οι κάτοικοι συγκεκριμένη χώρας να εργαστούν. Μιλήσαμε, αναφερθήκαμε για τη, στα δάση του Αμαζονίου και του ωκεανού, αλλά δεν μιλήσαμε για τα ευρωπαϊκά δάση. Ε, χρειάζεται διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείρισή του. Χρειάζεται ενημέρωση του κοινού ευρύτερη. Ε, Στου ε, πολίτε είναι δύσκολο να γνωρίζουν σήμερα πώ γίνεται η διαχείριση ιδιωτικού ή δημόσιου δάσου. Ε, αν θα υπάρξει πλήρη αποδάζωση ή καλύτερη διαχείριση. Άκουσα και την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής για τη νέα πράσινη συμφωνία, ρύθμιση για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των αρνητικών συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Το θέμα του δάσους είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού. Και εμείς εξακολουθούμε στην πόλη μου να αγοράζουμε διάφορα αγροτεμάχια για καλύτερη, πιο βιώσιμη εκμετάλλευση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιληφθεί καλύτερα αυτού του θέματος μαζί με τους ε, τοπικούς άρχοντες και να δούμε ε, το δάσος να θεωρηθεί ότι ήταν επένδυση και εξακολουθεί και θα εξακολουθεί να είναι επένδυση. Χρειαζόμαστε όμως μια βιώσιμη επένδυση και πρέπει να το αναλύσουμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ Βενσάν. να δώσω τη δυνατότητα σε δύο άλλα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών να εκφράσουν την άποψή τους, να μας πούν ποια είναι η εμπειρία τους και ίσως να θέσουν και κάποιο ερώτημα που θα απευθύνουν στα τρία εκπροσωπούμενα θεσμικά οργάνα. Και Φερνάντο Λόπες Μοιράς παρακαλούμε να σηκωθεί και να πει αυτό που θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ κατερχήν για αυτή την εναρκτήριο συνειδρίαση η οποία χαρακτηρίζεται από την νεότητα. Και πρέπει να πω ότι εγώ είμαι πιο νέος από το πόσες περιφέρειες έχει η χώρα μου. Αυτό θα πω μόνο. Και να σας πω πως για τη Μούρσια είμαστε στο νότο της ε, Ισπανίας και της Ευρώπης. Είμαστε εξαιρετικά τρωτοί λόγω κλιματικής αλλαγής γιατί προχωράει η ερημοποίηση η οποία θα καταλάβει και τη δική μας Ήπειρο αλλά δεν είναι η μοναδική απειλή. Επίσης οι νέοι δασμοί που επιβάλλουν η είναι μεγάλο χτύπημα για τη γεωργία μας ε, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τη Μούρσια μια και έχουμε σπεριδοειδή, ε, τυριά, κρασιά, λάδια και γι' αυτό ήθελα να πω πως η δική μου κυβέρνηση θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στεναρή στάση υπέρ όλων μας. Επίσης θα πρέπει να είναι στεναρή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πολιτική της κατά της κλιματικής αλλαγής. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς στο Νότο με την ερημοποίηση σύντομα θα φτάσει και στο κέντρο της Ευρώπης και στο Βορρά. Το φαινόμενο αυτό όπως ξέρετε προκάλεσε πριν από μερικές εβδομάδες φοβερές πλημμύρες στην περιοχή μας πρόσφατα. Πλημμύρες που έκαναν τις μεγαλύτερες ζημιές ποτέ σε σχέση ε, με τα στοιχεία που έχουμε από τη στιγμή που ξεκίνησε η καταγραφή στην Ισπανία. Ζητήσαμε βοήθεια λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους ζημιώθηκαν περισσότερο που ήταν κυρίως ο γεωργικός και ο τουριστικός κλάδος. Χρειαζόμαστε στήριξη. Στήριξη από αυτού με του οποίου μοιραζόμαστε τα κοινά ευρωπαϊκά μας σχέδια και θέλουμε να ενεργοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύας για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η φυσική καταστροφή και για να βοηθήσουμε ανθρώπους να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους το μέλλον τους γιατί οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι πάντα στο κέντρο και στον πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να παίξουμε στις πολιτικές που θα μας βοηθήσουν να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή και για το περιβάλλον και για την οικονομία και για τη χωροταξία και χρειαζόμαστε επίσης και είναι σημαντικό αυτό να έχουμε τις απαραίτητες υποδομές να μοιραστούμε τους πόρους με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε και απευθύνομαι σε εσά, Μέχρι πού θα φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει κατάλληλα και επαρκώς τη μάχη κατά της κλιματικής αγωγής έτσι ώστε να ε, μην προχωρήσει η ερημοποίηση και για να αποζημιώνονται όσοι έχουν ε, πληγεί από φυσικά φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή όπως η περιοχή μου πρόσφατα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τροφή προσκέψη. Τρίτο μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών. Παρακαλούμε να θέσει το ερώτημά του στους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση. Ο κ. Φρανκ Τσεκόνη, μέλος Επιτροπής των Περιφερειών από τη Γαλλία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ να σας πω πόσο χαίρομαι όπως και όλοι οι άλλοι που συμμετέχω σε αυτό το ραντεβού της Ευρώπης, της πραγματικής, είναι μια στιγμή που μα ενισχύει εμά, τα μέλη τη τοπική αυτοδιοίκηση, για να ολοκληρώσω αυτά που έλεγε ο Βανσάν. Δεν αμφισβητώ την ανάγκη να διαφυλάξουμε τα δάση. Είναι ουσιαστικό αυτό. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα έλεγα ότι χρειάζεται ένα σφαιρικό όραμα είναι το περιβάλλον με την αυστηρένεια του όρου, αλλά και οικονομικές παράμετροι και κοινωνικές πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σήμερα αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων ζει σε πόλεις και αυτή η τάση θα συνεχιστεί προφανώς μέχρι το 2050 και μετά από αυτό. Αυτό συνεπάγεται εντατικοποίηση της αστικοποίησης. Πάνω από τις ε, μισές πόλεις αντιμετωπίζουν τις ε, αρνητικές συνέπειες αλλαγής του κλίματος και απειλούνται ένα από τα μεγάλα προβλήματα να συμφιλώσουμε τους στόχου της μείωση της αλλαγής του, των αρνητικών συνεπειών τη αλλαγή του κλίματος στην πολιτική συνοχής. Γι' αυτό χρειάζεται προσαρμόγη. Η πολιτική τη συνοχής αύριο θα πρέπει απόλυτα να συνδράμει σε αυτή την προσαρμογή που τίνουμε να λησμονούμε. Τι τίθεται σε εμά σαν θέμα Όπω και έλεγε και ο Κριστιαν, αν προτιμούμε να ε, καθυστερήσουμε τι αλλαγέ, να πληρώσουμε το τίμημα ή να προβλέψουμε, να δραστηριοποιηθούμε έγκαιρα και να ελπίσουμε να συνεχίζουμε να ευημερούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε Μπιενκόφσκα, να σας ζητήσω να μείνετε πρώτοι. Ήδη απαντούσατε τις ερωτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα πριν, στην προηγούμενη παρέμβασή σας. Λοιπόν, η Επίτροπος, είμαι σίγουρη ότι αυτό που συζητούμε και που ξεκινήσαμε το συζητούμε από παλιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικό. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 θα είναι διαφορετικό από τα άλλα, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Φτάσαμε πολύ μακριά μέσω των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών προδιαγραφών και μέχρι τώρα και κατά τις προηγούμενες περιόδους της πολιτικής συνοχής είχαμε τρόπο να μειώσουμε τις εκπομπές οξυδίου του άνθρακος, να μειώσουμε τις σπατάλη ενέργειας, να αντιμετωπίσουμε την ε, ενεργειακή φτώχεια, να προσαρμοστούμε και να δημιουργήσουμε πράσινες υποδομές. Ήδη υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Και υλοποιείται αυτά τα προγράμματα, όπως ξέρετε. Ποια είναι η διαφορά τώρα, όπως προανέφερα. Το θέμα του κοινωνικού συναισθήματο που μας περιβάλλει διότι αισθάνεται ο κόσμος ότι είναι υπαριθμόν ένα θέμα για την Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά για την Ευρώπη είναι πολιτικά αποδεδειγμένο το πρώτο θέμα. Η κυρία Ούσολα Βόντερ Λάιεν το ανακοίνωσε άλλωστε ότι θα προτείνει αυτή την πράσινη ρύθμιση, το Green Deal, το πρώτο τρίμηνο της θητείας της. Αυτό είναι κάτι που θα είναι πρώτη στη μέρημνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια μέτρα, τι μέσα, τι πολιτικές, θα θεσπίσουμε στην Ευρώπη για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κοινωνικής στήριξης που υπάρχουν. Και για τους ανθρώπους, κυρίως τους νέους που τα περιμένουν αυτό. Θα έχουμε περίπου ένα 3 ευρώ επενδύσεις για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη. Και μεγάλα τμήματα της πολιτικής συνοχής θα υποστηρίζουν ε, αστικά προγράμματα η αστική ατζέντα θα ισχυροποιηθεί, διότι οι πόλει διαφορετικών μεγεθών, όχι μόνο οι μεγάλε πόλει, αλλά μεσαίου μεγέθου και μικρέ πόλει έχουν ανάγκε και ξέρουν πώ μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, την αλλαγή του κλίματο. Διαθέτουν τα μέσα τώρα. Και όπως ανέφερε κάποιος, έχουμε και το Ταμείο Μετάβασης που αφορά αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων αυτοί που θα αντιμετωπίσουν τα περισσότερα προβλήματα, τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιβαλλοντικής πτυχής μπορούν να προσφύγουν σε αυτό. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και με δίκιο τρόπο είναι τα χρήματα. Κάποιοι θεωρούν ότι το Ταμείο Μετάβασης θα είναι κάτι συμπληρωματικό πέρα από τον προπολογισμό μας. Ξέρετε σε ποιο κόσμο ζούμε. Θα έχουμε σύντομα το Brexit. Έχουμε ε, κράτη-μέλη που δεν θέλουν να πληρώσουν περισσότερα για να βάλουν στον ευρωπαϊκό κορβανά, τον κοινό κορβανά περισσότερα χρήματα. Το Ταμείο Μετάβαση θα είναι ένα από τα εργαλεία τη πολιτική συνοχή πιθανότατα. Δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα την πραγματικότητα. Δηλαδή, οι πολίτε μα θέλουν αυτή την πράσινη συμφωνία, το Green Deal. Θέλουν διαφορετική πολιτική λύση, θεσμική λύση για καθαρότερο ατμοσφαιρικό αέρα, για το κλίμα, για τα δάση, για το μέλλον του ανθρωπίνου είδους. Περί αυτού πρόκειται, αυτό συζητάμε. Από την άλλη, πρέπει να μοιραστούμε τους υπάρχοντες πόρους εφιός, διότι το επενδυτικό σχέδιο η πολιτική συνοχής με επίκεντρο της πόλης πρέπει να κινητοποιηθούν. Και έχουμε και το Ταμείο Μετάβαση για εκείνου που χρειάζονται περισσότερα μέσα, μεγαλύτερη υποστήριξη κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο. Ευχαριστώ, κυρία Μπιασκόφσκα. Πρόεδρε Λάμπερτ, εσεί τι πιστεύετε για το συγκεκριμένο θέμα τη ιωσιμότητα και τη αλλαγή του κλίματο. Θεωρώ ότι το μέλλον μας εξαρτάται από κάποιες βασικές Αλλαγέ που πρέπει να κάνουμε. Η αηφορία, η βιωσιμότητα, είναι καθοριστικής σημασίας. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε με τρόπο ευθύ. Πραγματικά ε, η φιλοδοξία της κυρίας Φόντερ Λάιεν να φτιάξει ένα πρόγραμμα σε 100 μέρες είναι εντυπωσιακό. Όμως η πολιτική μου εμπειρία τα τελευταία χρόνια μου έδειξε ότι όταν ορίζω τέτοιες προθεσμίες πρέπει να είμαι πολύ ε, επιφυλακτικός. Διότι δεν αρκεί να κάνουμε ένα πρόγραμμα, πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα σωστά εξορροπημένο και να μπορεί να λειτουργήσει. Και γι' αυτό πρέπει να συνδυαστούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ένα εξισορροπημένο πρόγραμμα Σημαίνει το να δούμε τι κοινωνικέ προεκτάσει ενό τέτοιου προγράμματο. Δεν ε, χρησιμεύει σε τίποτα μια περιβαλλοντική πολιτική μόνο ε, όταν μένει στα, στα λόγια και δεν μπορεί κανείς ε, στο τέλος του μήνα να βγάλει τα έξοδα. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία με τα κίτρινα γυλαίκα. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα έχουν άλλα θέματα και θέλουν την περιβαλλοντική διάσταση και την κοινωνική να τη λάβουμε ταυτόχρονα υπόψη και πρέπει να μπορέσουμε να του συμπαρασύρουμε όλου, ιδίω τι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι εκείνε πρέπει να υλοποιήσουν όσα αποφασίζονται στο επίπεδό του. Χρειάζονται και νομικά πρότυπα, αυτό μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά την πρακτική υλοποίηση την αναλαμβάνουν οι τοπικοί ηθήνοντε και οι περιφερειακοί δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα εάν δεν έχουμε αυτό το επίπεδο στο πλευρό μας. θα είναι μεγάλο κίνδυνος. Και βλέπουμε Επίσης τη διαφορετική πορεία, το διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης των αστικών κέντρων και το κέντρο της υπαίθρου. Ε, πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά το θέμα της συνεκτικότητας και της συνοχής στην Ευρώπη και πρέπει κυρίως να συγκεντρώσουμε αρκετούς πόρους. Ε, εκεί πολύ συχνά σταματάει η φιλία όταν φτάνουμε να μιλήσουμε για χρήμα. Ε, Όμω πρέπει να μιλήσουμε και για πόρου, διότι είμαστε μια από τι υπήρου από τι πλουσιότερε στον κόσμο. Τους, στα βιβλιάρια τα αποταμινιευτικά υπάρχουν και με αρνητικά επιτόκια δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κάτι το FES, να ε, κινητοποιήσουμε τους πολίτες, να διαθέσουν αυτά τα χρήματα ε, για την οικολογική ανανέωση της Υπήρου αλλά και με μια λογική κερδοφορία μπροστά τους για να έχουν κάτι να αποκομίσουν με αποτελέσματα ως προς την αηφορία. Εδώ λοιπόν έχουμε μεγάλο, πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να ξεκινήσουμε ως τα δυνατόν γρηγορότερα διότι είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για να πετύχουμε κάτι πολιτική της συνοχής. Ευχαριστούμε κυρία Λάμπερτς, κυρία Ντόμπρεφ. Ήδη μας σκεγγραφίσατε πώς θα τα δύο θέματα της βιωσιμότητας και της συνοχής. Νομίζω ότι από όλου μας τους ε, ομιλητές κάτι τέτοιο προκύπτει και είναι και πολύ σαφές. Ε, βεβαίως, Έχω σημειώσει τις ερωτήσεις σας. Το ερώτημα είναι θα είναι αρκετά ισχυρό το Κοινοβούλιο. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Συμβούλιο θα είναι και εκείνοι αρκετά τολμηροί. Κατάλαβαν πόσο σημαντικές αποφάσεις πρέπει να λάβουν τώρα, πόσο κέρυες και μάλιστα στο άμεσα προσεχές μέλλον, διότι δεν καταλαβαίνω ακριβώς την μεριμνά σας και αυτό είναι και το παράδοξο της δημοκρατικής πολιτικής. Βραχυπρόθεσμα η πολιτική εντολή είναι ένα πράγμα και μακροπρόθεσμα η παγκόσμια ανάπτυξη κάτι άλλο. Αυτό πάντοτε έρχεται σε αντιπαράθεση, σε αντίφαση και κάθε πολιτικός πρέπει να αντιμετωπίσει. Βεβαίω έχουν ακουστεί τόσες πολλές ανησυχίες για τις κλιματικές αλλαγές, όμως η πολιτική δεν ήταν έτοιμοι να λάβουν σκληρέ αποφάσει, αποφάσει για τι οποίε θα θυσίαζαν κάποιου μακροχρόνιου πολιτικού στόχου προσωπικού του ή τη βραχυπρόθεσμη πολιτική του εντολή. Εγώ όμω είμαι αισιόδοξη χωρί να είμαι αφιλή. Θέλω όμω να είμαι αισιόδοξη ότι κάτι κινείται στον κόσμο, ότι υπάρχει κάποια ε, μεταλλαγή στη στάση των πολιτικών. Εκατομμύρια νέοι κατεβαίνουν στους δρόμους σχεδόν κάθε Παρασκευή παντού στον κόσμο. Ε, η κοινή γνώμη, όπως θέλετε πείτε το, όπως σας αρέσει, είναι, φαίνεται να συγκινείται. Και πρέπει να πω κάτι στους φίλους ευρωβουλευτές και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Για ελάτε, για δείτε λιγάκι, αλλαγή χρειάζεται η κοντόφθαλμη πολιτική σας εντολή θα εξαρτηθεί από τι μακροχρόνιε πολιτικέ σα δεσμεύσει για τι κλιματικέ αλλαγέ. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξη για την ε, προσεχή λήψη αποφάσεων. Και βεβαίω δεν είναι εύκολο. Ναι, προφανώς τώρα το Κοινοβούλιο προτείνει την αναστολή προσφοράς βοήθειας από πόρους που πηγαίνουν για τα ορεκτά καύσιμα. Υπέροχο. Δεν μπορούσα παρά να συμφωνήσω περισσότερο. Όμως οι κεντρικές οι οικονομίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι περισσότερο εξαρτημένες από τον άνθρακα από ότι η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή η απαγόρευση λοιπόν πρώτον θα βαρύνει και θα πλήξει τι χώρε τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και έτσι ξαναπάμε στο πρώτο μα θέμα και την αλληλεγγύη. Διότι όταν λέμε πράσινη πολιτική, όταν λέμε καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, δεν μιλούμε μόνο για ηλιακούς κούς θερμοσύφωνες ή για δασοκομεία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όμως αυτό πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η αλλαγή στο σκηνικό δεν γίνεται μόνο στους δρόμους και τις διαδηλώσεις αλλά και στην πολιτική. Η πράσινη πολιτική είναι ιδιαίτερα περίπλοκη με μακροοικονομικές αλλαγές, συλλογιστική και προβληματισμό και μια νέα διάρθρωση, μια νέα διάρθρωση της κοινωνίας. Κάτι που σημαίνει μια νέα πράσινη οικολογική βιομηχανική πολιτική. Και το τονίζω πάντοτε μια ατζέντα, μια σειρά προτεραιοτήτων που να επιτρέπουν την κοινωνική συμμετοχή όλων. Διότι στο κάτω-κάτω τη γραφή από αυτόν τον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι μια ισχυρότερη, μια πιο ενωμένη Ευρώπη από ό,τι τώρα. Όπω σα είπα, είμαι αισιόδοξη χωρί να με θελεί. Είμαι αισιόδοξη, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι καθήκον έχουμε μπροστά μα. Ευχαριστούμε, κυρία Ντόμπρεφ. Πρέπει να επιστρέψουμε σε εσά. Θα περάσουμε λοιπόν στο slide.com για να απαντήσουμε και πάλι και θα ήθελα να μας πείτε εσείς τι πιστεύετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά φιλόδοξη στις δράσεις για το περιβάλλον. Ναι ή όχι. Ξεκάθαρη λοιπόν η αρχή. Αυτοί που ψήφισαν όχι ήταν πιο γρήγοροι, αλλά μοιάζει να εξισορροπεί. 60-40 λοιπόν, 60% από εσάς και από αυτούς που μας παρακολουθούν μέσω web streaming πιστεύουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει αρκετά και αυτό προκύπτει μάλλον από το γεγονός ότι εσείς κάνετε πολλά σε τοπικό επίπεδο αλλά αισθάνεστε πως στο θέμα αυτό χρειάζεστε στήριξη και για να γίνουν αυτά σε τοπικό επίπεδο θέλετε και οι πολίτες σας και οι εκλογικές σας περιφέρειες να ασχοληθούν περισσότερο. Πόσο λοιπόν ευαίσθητοι είναι οι πολίτες σας και πόσο γνωρίζουν τα όσα πόσο γνωρίζουν τα όσα γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς μπορούμε να σας φέρουμε πιο κοντά με αυτούς. Θα δώσω το λόγο στη Μία Σκαλίνα Φίγκερος που είναι τοπική σύμβουλος ε, στην Φιλανδία έχει αναλάβει ένα project στα πλαίσια μιας δράσης νέων ε, πολιτών για το για την πολιτική συνοχή, γιατί θέλετε να του δείξετε τι σημαίνει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και θα ήθελα, και θα ήθελα να σα ρωτήσω, πιστεύετε πω υπάρχει αρκετή αλληλεγγύη και πώς μπορούμε να φέρουμε τους Ευρωπαίους πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είμαι το ίδιο χαρούμενη όπως και η Λάουρα και θα δείτε τώρα τι σημαίνει ενθουσιώδης Φιλανδέζα αν συγκριθεί με ενθουσιώδης Ιταλίδα. Εν πάση περιπτώσει έχω ε, μαζί τα ε, σημειωμάτά μου και επειδή είμαι από την ε, Βόρεια Σλαβωνία, να σα πω ότι εμεί έχουμε μια παροιμία που λέει πω όταν κάποιο λέει κάτι, η ευθύνη βαρύνει αυτό που τον ακούει. Γι' αυτό λοιπόν τα έχω σημειώσει, γιατί είστε υπεύθυνοι εσεί. Να σα πω λοιπόν στο δικό μα project προσπαθούμε να βρούμε νέε καινοτόμε πλατφόρμε όπου ε, θα ενθαρρύνουμε του νέου να μπουν στη διαδικασία πολιτική διαδικασία λήψης απόφασης έτσι ώστε να ε, έχουν μια προσέγγιση η οποία θα είναι πιο θετική και να ρωτάνε τι θα γινόταν εάν εκτός ε, από τη συνηθισμένη πολιτική απάντηση η οποία είναι ναι μάλλον αλλά πάντως όχι. Επίσης πόσοι από εσάς έχουν γεννηθεί ε, που έχουν μετά το 1982 και μετά. Σηκώστε το χέρι σας. Εκεί πίσω κάθονται οι νέοι λοιπόν. Και μένα μου έκανε εντύπωση το ότι ανήκω σε αυτή τη γενιά, παρόλο που η Google λέει πως δεν μας αρέσει να μας αποκαλούν στα αγγλικά millennials. Να πω λοιπόν πως η δική μας ε, η δική μας κατανόηση του του είναι η συνοχή είναι μια φούσκα η οποία ή θα σκάσει ή θα παραμείνει. Οπότε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε οι πιο νέοι άνθρωποι να έρθουν κοντά μας στην ε, πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων και να καταλάβουν ότι με τον τρόπο αυτό ασκούν επιρροή. Να σας πω επίσης πως ο λαϊκισμός θα καταστρέψει την πολιτική μας δημοκρατία αν δεν καταφέρουμε να συνενώσουμε τον παλιό τρόπο που γινόντουσαν τα πράγματα με τον καινούριο. Η δημοκρατία ήταν σταθερή και αργή. Αλλά οι νέοι ζουν γρήγορα. Τα κοινωνικά δικτύα τα έχουν κάνει όλα πάρα πολύ γρήγορα. Η επικοινωνία έχει αλλάξει με ε, δραματικό τρόπο και θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο που θα συνδυάζει το παλιό με το καινούριο. Το σύστημά μας κινδυνεύει ε, να θεωρηθεί απαρχαιωμένο και να ατροφήσει γιατί οι νέοι θέλουν να επηρεάσουν, θέλουν να κάνουν αλλαγές Μιλάμε πολύ για το Green Deal εδώ. Ε, νομίζω ότι είναι πρωταρχικά θέμα νέων. Εμείς είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε το αύριο. Επίσης, είναι πολύ σχετικό το να ρωτάμε κατά πόσο η συνοχή, έτσι όπως εμείς την καταλαβαίνουμε, έχει κάποια σημασία για τους νέους. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουν οι ίδιοι πως είναι κομμάτι αυτού του σχεδίου που εμείς περιγράφουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να συνταχθούν μαζί μας και να ηγηθούν της δικής τους Ευρώπης και όχι αυτές τις οποίες χτίσαμε εμείς με τους δικούς μας κανόνες. Είναι καθήκον μας να ακούσουμε και να διευκολύνουμε την επικοινωνία και θα ήθελα ε, να σας παροτρύνω να σκεφτείτε ε, τελείως εκτός κανόνων. Μην μπείτε καθόλου στο πλαίσιο. Τι θα ήταν η Ευρωπαϊκή Συνοχή αν αποφάσιζαν οι νέοι. Αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε και αυτό θέλουμε να απαντήσουμε μέσω του project που έχουμε δημιουργήσει. Ευχαριστώ πολύ μία. Και τώρα θέλω να επιστρέψουμε σε κάποια από τα μέλη μας της Επιτροπή των Περιφερειών και να ακούσουμε κάποια σχόλια. Μετά θα ακούσουμε τα μέλη του πάνελ και μετά θα ξανακάνουμε τον κύκλο. Ο κύριος Ρομπ Γιούγκμαν από την Ολλανδία. Να εκφράσει τι απόψει του, παρακαλούμε. Ευχαριστώ, Φλόρενς. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή των Περιφερειών που σχημάτισε ένα τόσο ε, νεανικό ε, πάνελ με συμμετοχή τόσων νέων πολιτικών. Αν θέλουμε η Ευρώπη να πλησιάσει τους ε, πολίτες, είναι σημαντικό για μας να έχουμε ένα καλό πρόγραμμα, μια καλή ατζέντα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να καταρτήσουν τέτοιο θεματολόγιο. Θα πρέπει να περιγράφεται σωστά η κατάσταση, ξεκάθαρα, να θεσπιστεί μια νομοθεσία η οποία να είναι αυτή που καλύπτει τις ανάγκες. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει πάντα σε όλες τις λύσεις να περνάμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως και ο ελεύθερος ανταγωνισμός μπορεί να παίξει το ρόλο του. Μπορούμε να θέσουμε διάφορα ερωτήματα την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν υπάρχουν πολλά διοικητικά εμπόδια. Να δούμε αν υπάρχουν πολλά διοικητικά εμπόδια στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Θα πρέπει τελικά να, να δοθούν και δυνατότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ευρώπη είναι πολύ απόμακρη. Ε, θέλει να τα ρυθμίζει όλα από το κέντρο από τις ε, απόμακρες Βρυξέλλες. Αλλά, αλλά το τυρί, παραδείγματος χάρη, ε, το, ένα τοπικό τυρί που δεν εξάγεται θα πρέπει να το ρυθμίζει πώς παράγεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Θα πρέπει βασικά να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι λήψει αποφάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται στο πιο αποκεντρωμένο επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο δυνατόν, μετά περιφερειακό, μετά εθνικό και αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο τότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, είναι κάτι απαραίτητο για να πλησιάσει η Ευρώπη του πολίτε τη. Το πώ λειτουργούν τα θεσμικά όργανα τη Ευρώπη να αναλυθεί περαιτέρω. Θέλουμε να είμαστε εταίροι ε, η Επιτροπή των Περιφερειών. Η επιρροή τη τοπική αυτοδιοίκηση των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αρχών ε, είναι κάτι που δημιουργεί την εμπιστοσύνη. Να μην είσαστε εδώ σε έναν χρυσελεφάντινο πύργο στις Βρυξέλλες, αλλά στο Κατόβιτσε, στη Φλωρεντία, σε οποιαδήποτε πόλη, στη Βαρσοβία, οπουδήποτε, ε, να αισθάνονται ότι το, μπορούν να βρουν τις λύσεις. Να πλησιάσει η Ευρώπη, ε, τους πολίτες πώς θα εφαρμόσετε την επικουρικότητα και να είσαστε πιο κοντά στους ε, πολίτες εάν δεν κινηθείτε προς την αποκέντρωση. Να λαμβάνονται υποφάσεις κοντά στον πολίτη. Ευχαριστώ κύριε Γιόγκμαν. Λοιπόν, ε, προχωρήσαμε προς διαφορετικό θέμα, κινηθήκαμε προς την επικουρικότητα. Ε, αλλά είναι κάτι που έχει αντίκτυπο. Οι εθνικές αποφάσεις καμιά φορά και αυτές μπορούν να επηρεάσουν την Ένωση. Θα ήθελα τώρα να στραφώ προς το τελευταίο μέλος του πάνελ, την Κριστίν ε, Κάρι, που είναι μέλος του Highland Council του Ηνωμένου Βασιλείου και μαντεύεται για τι πράγματα μιλήσουμε. Η Κέρστιν, Κέρστιν μάλλον πριν από τρία χρόνια, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισαν να ψηφίσουν υπέρ του Brexit. Παρότι ξέρουμε ότι η Σκοτία δεν ψήφισε υπέρ του Brexit, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει κάποιες ευθύνες όσον αφορά το αποτέλεσμα της ψήφου. Τι χάσαμε, πού κάναμε λάθος όσον αφορά την επικοινωνία μας με τους πολίτες. Πώς μπορούσαμε να τους ε, αφήσουμε να, να φύγουν παρά να τους ενημερώσουμε να τους κρατήσουμε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα πολύ. Μίλησα στα γοδελικά την τοπική γλώσσα της Σκωτία. Όχι μόνο έχουμε την τοπική μας διάλεκτο, την τοπική μας γλώσσα, αλλά ψηφίσαμε διαφορετικά στη Σκωτία και θέλαμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Δυστυχώς το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ξέρουμε, δεν ψήφισε να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για μένα νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά τον ανεξέλεγκτο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης που έχουν επί των πολιτών μας και τα μηνύματα που έβγαιναν από το ΜΜΕ. Ε, μηνύματα λαϊκισμού έβγαιναν. Όπως ακούσαμε και πριν, αυτό είναι κάτι τρομακτικό, φρικτή κατάσταση. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες της Σκωτίας επηρεάζονται λιγότερα από το ΜΜΕ. Ε, νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί στη Σκωτία από το 1999 ε, Εξανάρχισε τη λειτουργία του το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο και είχαμε κυρίω κυβερνήσεις αριστερές, κέντρο αριστερές που πρόβαλαν θετικό, ε, θετική εικόνα θετική αντιμετώπιση ε, των θεμάτων των ε, κοινωνικών, των οικονομικών και της κοινωνική συνοχή περιθωριοποιημένε κοινότητε στη Σκωτία αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται περισσότερο από ό,τι αντίστοιχε στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Χάρη μεταξύ άλλων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οπότε έρχομαι σε αυτό που είπε Φλόρεν. Τι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε κάνει καλύτερα. Όλε οι κυβερνήσει, πιστεύω σε κάθε επίπεδο πρέπει να κινηθούν ε, και να έρχονται σε επαφή με διαφορετικό τρόπο με του πολίτε. Οι παλιοί τρόποι επαφή δεν λειτουργούν πια και ε, έχουμε επικρατεί το χρήμα και τα τρομακτικά μηνύματα και πρέπει να βρούμε καινοτόμους τρόπους, πραγματιστικούς τρόπους για να περνάμε τα μηνύματά μας στους πολίτες, να τους δείξουμε τι σημαίνει να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ρωτήσω οποιονδήποτε δεν ξέρει κανείς τίποτα από, τον απλό, από τους απλούς ανθρώπους για την πολιτική συνοχή ή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δεν είναι κάτι που εξηγείται στους απλούς πολίτες, δεν αισθάνονται συμμετέχουν, αισθάνονται περιθωριοποιημένοι. Ποια είναι η πραγματικότητα κατά την άποψή μου. Πρέπει να πλησιάσουμε τους ευάλωτους ανθρώπους σε όλες μας τις κοινωνίες και να τους φέρουμε μαζί μας το ταξίδι που κάνουμε, να μιλήσουμε στον κόσμο, να τους κάνουμε να καταλάβουν, να κατανοήσουν Πώς συμμετέχουν στο, στην εικόνα αυτή τη ψηφιδωτό που δημιουργείται, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορα κομματάκια, που ανήκουν και αυτοί σε αυτή την εικόνα. Ευχαριστώ πολύ, Κριστίν. Και μια τελευταία παρέμβαση από τους ομιλητές μας. Από τους προσκεκλημένους μας μάλλον. Ο κύριος Καν Βον Λόουερ. Ευχαριστώ. Στα Ολλανδικά κι εγώ. Κυρίε και κύριοι προσκεκλημένοι νέοι πολιτικοί, ακούσαμε μια σειρά από ενδιαφέρουσες δηλώσεις. Έχουμε εδώ ηγέτες του μέλλοντος. και όπως και εμείς εργάζεστε σε τοπικό επίπεδο, πιο κοντά στους πολίτες, πιο κοντά στους ψηφοφόρους. Γνωρίζετε τι συμβαίνει στην πράξη. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νέο Ευρωκοινοβούλιο χρειάζονται μια πιο σφαιρική προσέγγιση για να συμμετέχουν περισσότερο οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης και οι ίδιοι πολίτες. Χρειάζεται λοιπόν μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Όχι να, να επιβάλλουμε τις πολιτικές αποφάσεις ε, άνωθεν, αλλά αντιστρόφως να ξεκινάει η χάραξη πολιτικών από τους πολίτες πολλά μέλη του Κοινοβουλίου, πολλοί επίτροποι. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησαν την καριέρα τους από τις τοπικές ε, πολιτικές διαδικασίες. Και στην ομάδα εργασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει την σημασία της αρχής της επικουρικότητας που θα πρέπει να διατρέχει και να διαπερνά εγκάρσια όλε τι πολιτικέ. Σε τι επίπεδο δηλαδή πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσει για τι κοινωνικέ πτυχέ, για τα θέματα πολιτισμού, για τα εκπαιδευτικά. Την περασμένη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, σε μια από τι ακροάσει συγκεκριμένα του κυρίου Σεύκοβιτ, ακροάσει των ε, υποψήφιων Ευρωπαίων Επιτρόπων, ο κ. Σεύτσοβιτ ε, ξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τον τρόπο που εργάζεται η Επιτροπή των Περιφερειών. Και εγώ θέλω να πω ότι ήταν πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε σε συνεργασία με περιφερειακέ και τοπικέ κυβερνήσει. Η ερώτησή μου λοιπόν σήμερα είναι πώ φαίνεται να διαμορφώνεται το μέλλον για την ε, επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον, το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Πώ σκοπεύετε να συνεργαστείτε με τοπικέ και περιφερειακέ κυβερνήσει για να βελτιωθεί η υλοποίηση μέτρων για την επικουρικότητα σε όλα τα επίπεδα. Και πώς θα γίνει αυτό σε περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς όπως η δική μου περιοχή, η Φλάνδρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Φάντεν Λόι. Να ακούσουμε τώρα τους θεσμικούς μας εκπροσώπους. Ακούσατε τις παρατηρήσεις, ακούσατε τις ερωτήσεις. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν δυσκολίες μέχρι να ε, μπορέσουμε να αγγίξουμε τους πολίτες. Υπήρχε το θέμα της επικουρικότητας. Κύριε Λάμπερτ, στην Επιτροπή των Περιφέρων, κατά την άποψή σας, πώς επηρεάζει αυτά τα πράγματα. Εάν έπρεπε να ορίσουμε την Επιτροπή των Περιφερειών, πιστεύω ότι δύο πράγματα θα έπρεπε να πούμε ότι είναι μέρος που τα συμβολίζουν. Πρώτα απ' όλα η συνοχή και μετά η επικουρικότητα. Η επικουρικότητα, αυτή η πολύ παλιά έννοια η σύλληψη ε, ότι πρέπει να λαμβάνονται αποφάσει στο επίπεδο που είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερο στου πολίτε και να συμμετέχουν οι πολίτε όσο το δυνατόν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων είναι μια αρχή ε, πολύ σημαντική. Και αυτό αν θέλουμε τα πράγματα να αλλάξουν στην Ευρώπη Είναι σημαντικό. Η Ευρώπη είχε πολλές φορές την τάση να ρυθμίζει διάφορες υποθέσεις και καταστάσεις καταλεπτός με μεγάλη επιμονή στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε τι πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εθνικό και μετά σε επίπεδο αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά κυρίως πρέπει να αναρωτηθούμε επίσης με τι συχνότητα, με τι πυκνότητα πρέπει να αποφασίζονται, να λαμβάνονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλέ φορέ είναι καλύτερα αποφάσει να λαμβάνονται κατευθείαν από τι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί που ο κόσμο ξέρει τι συμβαίνει στην πράξη. Πριν από λίγε μέρε είχα συνομιλία με, με την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Φόντερ Λάιεν, και εντυπωσιάστηκα. Εντυπωσιάστηκα το γεγονό ότι αυθορμήτω μου είπε τι εμπειρία είχε η ίδια από ε, την εμπειρία της ως Δημοτική Σύμβουλος σε μια μικρή πόλη στην κάτω Σαξονία και ως τοπική υπουργό στο κρατήδιο αυτό της Γερμανίας. Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε και μάλιστα στην ομιλία τη στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του στο Στρασβούργο, μίλησε για την ιδιαίτερη σημασία των αρχών τοπική αυτοδιοίκηση στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι η επικουρικότητα πραγματικά είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Και χαίρομαι που και στην προηγούμενη θητεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορέσαμε στην ομάδα δράση για την επικουρικότητα να εργαστούμε επισταμένω επί του θέματο. Αντλήσαμε κάποια διδάγματα και αναπτύξαμε μία έννοια της ε, ενεργούς επικουρικότητας. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό παιχνίδι, λες και ρίχνουμε πασχέτζα ή παίζουμε μια τράπουλα. Όχι, ε, είναι ένα θέμα ε, κέρια σημασίας και θα είναι μεγάλη επιτυχία εάν μπορέσουμε στην επικουρικότητα να συμπαρασύρουμε και τις αρχές τοπικές αυτοδίκησης στον ίδιο σκοπό, στον ίδιο στόχο. Ε, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαδικασία των τριμερών διαλόγων και εκεί να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρχών τοπικής αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι που ενθουσιάζει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αλλά το να μιλάμε για επικουρικότητα και να αποφασίζεται αυτό από δύο θεσμικά όργανα όταν ε, κάνει μια νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκεί. Πρέπει να συμμετέχουν και οι τοπικοί λειτουργοί. Ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρε Ντόμπρεφ. Πολλά τα ερωτήματα περιορισμένος ο χρόνος θα σας ε, επιβεβαιώσω πως εγώ θα είμαι πραγματικός εταίρος έτσι ώστε να έχουμε δυνατά τοπικά και περιφερειακά προγράμματα και όπως είπα και ε, πριν θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κονδύλια να έρθουν όσο πιο κοντά μπορούν στους πολίτες. Επειδή όμως υπάρχει περιορισμός χρονικός θέλω να μιλήσω για την επικοινωνία και μιλάμε και για τον Brexit θα αυτά. Λοιπόν, θα πρέπει παγκόσμια και από κοινού θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές του κλίματος. Ναι, αλλά έχουμε και μια πολύ μεγάλη απειλή που κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας που είναι η παραπληροφόρηση, τα, οι ειδήσει, τα fake news και εγώ είμαι από την Ουγγαρία, ψηφίσ... Ε, ξέρω τι σημαίνει fake news και τώρα με τον Brexit βλέπουμε πάρα πολλά αντίστοιχα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο ισχυρά εργαλεία για να δώσουμε τη μάχη κατά της παραπληροφόρησης και των fake news. Θα ήθελα η νέα θητεία του Κοινοβουλίου και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηριχθούν σε πολιτικό επίπεδο περισσότερο έτσι ώστε να δώσουν τη μάχη κατά αυτών των φαινομένων. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι καταρχήν μία πολιτική φύση επικοινωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεύτερον μεγάλες προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο. Εσείς είστε πολύ πιο πιστευτοί από αυτούς που κάθονται στο Στρασβούργο στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα κοινό θεματολόγιο, ένα κοινό σχέδιο μαζί με τα ε, εκατομμύρια ερετούς οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις στην Ευρώπη για να δούμε τι θα κάνουμε γιατί αφενός θα ήθελα να σας παροτρύνω και είμαι πολύ ικανοποιημένη που έχουμε προγράμματα για τους νέους έτσι ώστε να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε να επικοινωνούν, έτσι ώστε να εμπλακούν στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα. Τα στοιχεία από το Brexit. Οι δεν παρασύρθηκαν από τα fake news. Ψήφισαν υπέρ της Ευρώπης ως πλειοψηφία. Οι ηλικιωμένοι, αυτοί που ζουν στην Ήπεθρο, επηρεάστηκαν περισσότερο από τα κοινωνικά δίκτυα και από τα άλλα εργαλεία με τις ψευδείς ειδήσει και με τη διασπορά αυτών. Να κάνουμε λοιπόν μια εκστρατεία για τους νέους και να τους πούμε δίδαξε τον παππού και τη γιαγιά και τους γονείς ποιον εμπιστεύονται και ποιον όχι γιατί αυτό που βλέπω είναι πως οι νέοι κάνουν τη διαφορά πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουν οι πιο ηλικιωμένοι. Άρα λοιπόν το δεύτερο κοινό μας καθήκον σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο είναι να κάνουμε μια προσπάθεια να πατάξουμε τα fake news και την παραπληροφόρηση για να καταστρέψει τις χώρες μας και πιστέψτε με, ξέρω γιατί μιλάω. Σίγουρα λοιπόν μια αποστολή για όσους γεννήθηκαν μετά το 82. Κυρία Μπιανκόφσκα, σίγουρα για αυτούς γιατί όπως άκουσα με μεγάλη χαρά το καθήκον μας είναι να επικοινωνούμε. Και αυτό είναι αλήθεια. Η επικοινωνία και θα μιλήσω πρώτα για την επικοινωνία και μετά για την επικουρικότητα. Η επικοινωνία λοιπόν είναι δική μας ευθύνη σε άλλα επίπεδα. Ξέρω πως όλοι αυτή τη στιγμή λένε ναι οι ευρωβουλευτές, ναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς δεν τα πήγαμε άσχημα τα τελευταία πέντε χρόνια. Εκατοντάδες συναντήσεις ε, με τους πολίτες. Εγώ προσωπικά σε τουλάχιστον 100 ε, τέτοιες συναντήσεις ε, στις μικρές κοινωνίες παντού στην Ευρώπη για να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία είναι ευθύνη δική μας και επίκαιρα. Και επειδή μιλάμε για την επικοινωνία, έχουμε ψευδείς ειδήσει, έχουμε fake news και χρειάζεται ίσως σχετική νομοθεσία. Έχουμε τη βάση έτσι ώστε να εργαστεί το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κόσμος γύρω μας αλλάζει πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν και γι' αυτό προσπαθούμε και τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και συζητάμε κάτι το οποίο είναι πρόβλημα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήθελε στην προηγούμενη πενταετία να ε, παρουσιάζει συνέχεια καινούργια νομοθεσία, να μην προσθέτουμε νομοθεσία στην υπάρχουσα. Είχαμε αυτό τον κανόνα, το είπε και η κυρία Φαντερ Λάγεν που είναι μία νομοθεσία σε ισχύ, μία καταργείται, αλλά νομίζω ότι και ε, στην ε, ενιαία αγορά θα πρέπει να έχουμε τον κανόνα που θα είναι μία καινούρια ρύθμιση εισάγεται, 27 καταργούνται για να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών. Και ξέρω γιατί μιλάω. Κανείς δεν μπορεί να με καταγορήσει ότι ε, μου αρέσει να λειτουργώ σε κεντρικό επίπεδο γιατί εγώ αποκέντρωσα ε, τα ευρωπαϊκά ταμεία στην Πολωνία και τα περισσότερα κονδύλια πηγαίνουν κατευθείαν στις περιφέρειες. Ελπίζω να αλλάξει αυτό στο μέλλον, αλλά είναι κάτι που έκανα. Και έτσι λειτουργούν καλύτερα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι περιφερειακές, οι τοπικές αρχές, κάθε μικρή πόλη και χωριό. Εσείς είστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Εσείς πρέπει να επικοινωνείτε γιατί είναι μια αλυσίδα Μια αλυσίδα που μέσω τέτοιων εκδηλώσεων καταφέρνουμε να καταλάβουμε ποιες είναι πραγματικά οι προτεραιότητες, προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν και πώς θα παρθούν οι αποφάσεις στις Βρυξέλλες και θα εφαρμοστούν αλλού. Εγώ είμαι από την περιφέρειά μου, εγώ είμαι από τη μικρή μου πόλη. Ξέρω πως οι αποφάσεις των Βρυξελών είναι μακριά από εμάς και εσείς είστε τα σημεία επαφής και εσείς μπορείτε να μεταδώσετε και να εξηγήσετε τις αποφάσεις αυτές στους πολίτες. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και ξέρω πως η μελλοντική επιτροπή δεν θέλει καθόλου ε, κεντρική διαχείριση από τις Βρυξέλλες. Είμαστε διαφορετικές χώρες, διαφορετικές περιφέρειες, διαφορετικοί πολίτες, διαφορετικά χωριά. Ε, αυτή είναι η ομορφιά της Ευρώπης και είναι κάτι το οποίο μας κρατάει μαζί. Τι είναι, οι αξίες μας, η αλληλεγγύη, η πολιτική συνοχής. Έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο είναι κοινό μας και θα πρέπει όλοι αυτό να το κοινωνήσουμε στους πολίτες μας. Ξέρω πως ε, ε, ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι πριν από 5-10 χρόνια γιατί μας επιτίθονται από πάρα πολλές πλευρές και δεν γνωρίζουμε δεν ξέρουμε τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Είναι όμως δική μας ευθύνη. Και η επικουρικότητα είναι κάτι που θα τα πετύχετε εσείς, γιατί εσείς γνωρίζετε τις τοπικές σας κοινωνίες, τους τοπικούς σας πληθυσμούς. Κανείς δεν τα ξέρει καλύτερα. Εσείς και μόνο εσείς. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Η εθνική λήψη αποφάσεων περνά από τι εθνικέ κυβερνήσει, αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι εσεί δεν τα γνωρίζετε, γιατί δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική συνοχή και δεν μπορεί να εφαρμοστεί κεντρικά. Time to hear what... Ευχαριστώ, Επίτροπε Μπιανκόφσκα. ακούσουμε εσείς τι σκέφτεστε. Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση. Ξανά στο Slido πάμε. Slido.com Ποιος είναι σε καλύτερη θέση να επικοινωνήσει με τους πολίτες, να προωθήσει την επαφή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών. Ποιος μόνο το καταφέρει καλύτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις. Γρήγορη απάντηση βλέπουμε εδώ. Κοινωνία των πολιτών, άλλοι Αναφέρθηκαν τα μέσα ενημέρωσης Φερρυπίν. Αν περιμένουμε κι άλλο, δεν θα υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, πιο πολύ τονίσατε τους αυτούς σας. Βάλατε το βάρος επάνω σας. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ελπίζω να έχετε το υλικό στα χέρια σας, να αποκτήσετε το υλικό για να εκπληρώσετε την αποστολή σας που μόλις αναλάβατε. Διότι αυτό κάνατε, αναλάβατε μια αποστολή. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να δώσω ένα λεπτό σε κάθε έναν από τους ομιλητές μας για τελικά σχόλια περί των συζητηθέντων, περί των παρατηρηθέντων τι υπενθυμίσεις μπορούμε να κρατήσουμε από τη συζήτηση. Η Κριστίν. Πιστεύω ότι όλα αυτά που συζητούσαμε το απόγευμα μας πηγαίνουν στην έννοια της ελπίδας. Πολλοί πολίτες στην Ευρώπη, κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως στη Σκοτία δεν αισθάνονται ότι υπάρχει ελπίδα τώρα. Είναι ευθύνη όλων μας να ξαναδώσουμε ένα μήνυμα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης φιλίας, αγάπης ως ηγέτες να το μεταδώσουμε στις περιφερειές μας να στείλουμε ένα καλύτερο, πιο θετικό αφήγημα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βανσάν, εσύ τι αποκόμισες από τη συζήτηση. Να απαντήσω λίγο σε αυτά που υπόθηκαν σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Να χρησιμοποιήσουμε το πρίσμα των πόλεων. Η αστικοποίηση συνεχίζεται στην Ευρώπη, αλλά η ο πληθυσμό. Υπάρχει πληθυσμό ακόμα στην Ήπεθρο. Μιλήσαμε για το Brexit πριν. Στην Ήπεθρο κερδίζει έδαφο ταχύτερα ο λαϊκισμό. Η Ήπεθρο καταψήφισε την Ευρώπη. Στη Γαλλία υπάρχει ε, μια ταινία που αναφέρεται στην ιστορία της αυτοκτονίας ενός ε, Γεωργού ε, και αυτή η πολιτική συνοχή της μετάβασης ενεργειακής, η κοινωνική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ε, την, ε, τα συναισθήματα που επικρατούν, δυσαρέσκεια επικρατεί στην Ήπεθρο, που είναι το κλειδί για τη λύση, για τη μετάβαση και την προστασία του κλίματος. Να πω σε εκείνους που μας παρακολουθούσαν από το διαδίκτυο και τους εθνικούς βουλευτές και τους βουλευτές εν γέννη, ότι δεν αναφέραμε ε, τους πολιτικούς μας τίτλους, πολιτικές ιδιότητες. Αυτό το υποδεικνύει ότι στα δημοτικά συμβούλια ε, δεν είμαστε καν μέλη του πολιτικού κόμματος. Άρα δεν έρχεται μέσα πολιτική αντιπαράθεση η λύση, αλλά από ένα κοινωνικό μοντέλο, όπως είπε ο πρόεδρος Λάμπερτς. Τι θέλουμε να κάνουμε πρέπει να δείξουμε. Από εκεί βγαίνει η λύση και τη δυνατότητα να κινηθούμε ομαδικά για να βρούμε γρήγορα λύσεις και να βρούμε και τα χρήματα, τα αναγκαία για να πετύχουμε τους στόχους και τις λύσεις. Αντιπρόεδρε Ντόμπρεφ, εσείς τι έχετε να πείτε. Να σας πω. Μια σύντομη ιστορία Είχα καθηγητή στον πολιτικών επιστημών παλιά στο Πανεπιστήμιο και μου έλεγε ότι υπάρχουν δύο είδη πολιτικών. Ένα είδος είναι η αφηρημένη πολιτική. Κάθονται στα κοινοβούλια. Και μετά υπάρχουν αυτοί που πατάνε τα πόδια του στο έδαφο, αυτοί που είναι στα, στους δήμους. Οι πραγματικοί πολιτικοί που συναντούν τον άνθρωπο καθημερινά βρίσκουν τον απλό άνθρωπο. Αυτοί στο κοινοβούλιο ασχολούνται με αφηρημένου αριθμού, στοιχεία και νομοθεσία. Νομίζω ότι σε αυτή την ε, περίπτωση ήταν και θέμα προτίμησης. Καταλαβαίνετε αμέσως ποιον προτιμούσε ο καθηγητής μου. Αλλά από την πλευρά μου να σας πω ότι σαν αντιπρόδοση υπεύθυνη για την Επιτροπή των Περιφερειών και τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα έχετε ένα πολύ ισχυρό εταίρο, σας διαβεβαιώνω. Ε, είμαι σίγουρη ότι μια καλή ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τη συνεισφορά, την εποπτεία ε, των πιο ε, πρακτικών πολιτικών που ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Να αισθάνεστε ελεύθεροι, να έρχεστε σε μένα, ε, να εκφράζεστε ελεύθερα, να διαμαρτύρεστε αν κάτι δεν πάει καλά και εγώ θα προσπαθήσω να βρω τη λύση και διορθώσω. Ευχαριστούμε. Μία. Ναι, νομίζω ένα από τα καλύτερα που έγιναν σήμερα είναι ότι βρισκόμαστε εδώ καθισμένοι στην καρδιά, για να το πω έτσι, της Ευρώπης, αλλά το μήνυμα είναι, δεν είναι η καρδιά της Ευρώπης εδώ από μόνη της. Εμείς τη φέραμε. Εμείς κάνουμε την Ευρώπη αυτό που είναι. Και η δική μας απάντηση θα την κάνει ένα καλύτερο τόπο για να ζει κανείς. Να επικοινωνούμε καλύτερα και να προσαρμοζόμαστε σε αυτά τα προγράμματα που επιτρέπουν τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας. Έτσι θα γίνουμε δυνατότεροι. Ευχαριστούμε Ράντοσλαβ. Εσύ τι έχεις να πεις για όλη αυτή τη συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της εβδομάδας των περιφερειών και των πόλεων διότι έτσι έχουμε μια πλατφόρμα ως τοπική ηθήνοντες για να εκφράσουμε τη γνώμη μας. Είναι σημαντικό διότι θα πρέπει να μας υπολογίζουν τα θεσμικά όργανα και να τους απασχολεί το τι έχουμε να πούμε. Πρέπει να βρούμε ένα καλό σημείο ισορροπίας για το τι χρειάζεται να φέρει η νομοθεσία προς το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και έτσι να μετατρέψουμε την Ένωση των 27 κρατών μελών όχι σε έναν οργανισμό ομοιογένειας και όπου όλα θα είναι πανομοιότυπα αλλά η ποικιλομορφία να έχει τη θέση της. Ευχαριστούμε Επίτροπη Μπιενκόφσκα το δικό σας το συμπέρασμα. Πιστεύω εκβαθέων ότι η εσωτερική αγορά στην Ευρώπη χρειάζεται πολύ συνοχή. Και κατά τον ίδιο τρόπο η Ευρώπη συνολικά χρειάζεται ισχυρές περιφέρειες, ισχυρές πόλεις και ισχυρές τοπικές κυβερνήσεις. Αυτή είναι και η ομορφιά της Ευρώπης. Γι' αυτό και το συζητάμε σε μια τέτοια εκδήλωση και ξέχασα στην προηγούμενη παρέμβασή μου να πω ότι είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία των, της Επιτροπής των Περιφερειών που λέγεται RAPAP για να συζητήσουμε με πόλεις, περιφέρειες, τοπικές κυβερνήσεις τι κάνουμε πραγματικά. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία χρειάζεται πραγματικά στην πράξη. Και έχει ήδη προσφέρει πολλά ακόμα και κάποιες εκθέσεις εκπονήθηκαν. Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να συζητήσουμε το μέλλον μας τις δραστηριότητες της μελλοντική Επιτροπής για πολλά ζητήματα. Η τρίτη μου η παρατήρηση είναι ότι εσείς είστε η Ευρώπη. Πραγματικά εσείς είστε. Εσείς πρέπει να έρθετε σε επαφή, σε επικοινωνία με τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι μεγάλη η ευθύνη σας. Κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει μια Ευρώπη που δεν διέπεται από ποικιλομορφία. Κανείς δεν θέλει μια Ευρώπη που να είναι ομοιογενής Θέλουμε την Ευρώπη με αυτή την ομορφιά που διαθέτουν οι διαφορετικές της περιφέρειες, πόλεις. Χρειαζόμαστε διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να τα συζητήσουμε. Αλλά με μια κοινή αντίληψη, κοινέ ιδέες. Θέλουμε να είμαστε μαζί και να συνεπάρχουμε. Θέλουμε να είμαστε μαζί, θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή την Ένωση με όλη μας την ποικιλομορφία. Και αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους που γεννήθηκαν γύρω στο 2000. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και παραδείγματα ωραία όπως το Εράσμους και να εξηγήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη να την κατανοήσουν για να έρθουν όλοι πιο κοντά μας. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Μπιενκόφσκα. Λάουρα, εσύ ξεκίνησες. Ας κλείσουμε τώρα τον κύκλο. Πριν δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο Λάμπερτ. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε τώρα. Εμάς, η ποικιλομορφία μας είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, πιστεύω πως αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις. Προκλήσεις που θα αλλάξουν τον κόσμο. Όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας. Δεν γνωρίζουμε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα και ξέρουμε πως ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα, θα είναι πάντως διαφορετικά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο δυνατοί, πιο θαραλέοι. Θα πρέπει δηλαδή να δρούμε σε τοπικό επίπεδο, αλλά να σκεφτόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και πρέπει να είμαστε πιο συνδεδεμένοι μεταξύ μας πιο δικτυωμένη, Άρα το κοινωνικό σύστημα θα πρέπει να αλλάξει. Το κοινωνικό σύστημα δεν είναι ε, κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά έχει να κάνει με ελάχιστο βασικό μισθό, ε, έχει να κάνει με ε, παιδεία, με ευκαιρίες, με απασχόληση με επαγγελματικό προσανατολισμό. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που για κάθε άνθρωπο που είναι κάτω από τα 30 θα έχουμε και τρεις που θα είναι πάνω από τα 85. Θα είμαστε πάρα πάρα πολύ γέροι. Αυτό είναι καλό ότι σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή ποιότητα ζωής, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε οπτική γωνία και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και δεν είναι αν θέλουμε, επειδή θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να συζητάμε νέα κοινωνικά συστήματα και χαίρομαι που σχεδόν όλοι μας ε, μοιραζόμαστε αυτή τη σκέψη, ίσως από άλλη οπτική γωνία Είμαστε λοιπόν η καρδιά και τα χέρια. Αν εμείς, εμείς οι περιφέρειες, οι τοπικές κοινότητες, οι πόλεις, είμαστε τα χέρια τα οποία συνδέονται με την καρδιά που βρίσκεται εδώ και με το μυαλό που είναι ακόμα εδώ, τότε θα τα πάμε καλά. Αν κάποιος από μας δεν συνδέεται, θα καταρρεύσουμε. Και δεν είναι αυτό που επιθυμούμε. Παρακαλώ λοιπόν θα πρέπει τον άνθρωπο, να το βάλουμε στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιστρέψουμε σε αυτό που ήμασταν και να βρούμε αυτό που θα γίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λάουρα. Πρόεδρε Λάμπρετς. Υπάρχει ένας απλός τρόπος να συνοψίσουμε τα όσα συζητήθηκαν γιατί είμαι περισσότερο από ποτέ Πώ πως δεν είναι Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Στρασβούργο ή Ευρώπη, παρόλο που είναι όμορφες πόλεις. Η πραγματική ειναι ομορφες πόλει. είναι εκεί που ζει ο κόσμο, στι μικρέ τοπικέ κοινωνίε, στα χωριά, στις πόλεις, περιφέρειες και εκεί θα πρέπει να του πείσουμε και στο μυαλό και στο στομάχι και στην καρδιά πως θα συνεργαστούμε για την Ευρώπη γιατί αυτό δίνει μια προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και αυτή είναι η πρόκληση την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες οι γενιές. Με αποφασιστικότητα και με θέληση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, νομίζω πως ήταν πολύ ε, φορτισμένη και έντονη η συζήτηση και το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ελπίζω πως έτσι θα συνεχίσει και εύχομαι να περάσετε μια πολύ ε, ενδιαφέρουσα εβδομάδα, να μιλήσετε πολύ μεταξύ σας, να βρείτε δράσεις και σας παρακαλώ πολύ ας ευχαριστήσουμε το πάνελ με ένα χειροκρότημα. we please thank also the interpreters because they've had quite a bit of work to do thank you ladies and gentlemen and our technical team without whom that wouldn't be possible so thank you folks there is a bus waiting outside Έχει ένα λεωφορείο έξω στην πλατεία του Λουξεμβούργου για να πάτε όσοι θέλετε στην ξενάγηση για το επόμενο τμήμα αυτού του απογεύματος. Από ό,τι ξέρω έχουμε μια βραδιά γευσηγνωσίας. Στην πλατεία του Λουξεμβούργου είναι το ραντεβού στα λεωφορεία και βγαίνοντα, μην ξεχνάτε να κοιτάξετε και το βίντεο μα ε, τη εβδομάδα για τι Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.